ψηφίσουμε την Πέμπτη. Περνάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσια διάταξης που είναι οι παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Θα αρχίσουμε τον κύριο Χέις για ένα λεπτό. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να αποτανθώ στο σώμα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα του ε, ε, λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάνονται 10 δις ευρώ ετησίως και το 11% των τσιγάρων που πολλούνται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράνομα. Στην Ελλανδία το ποσό αυτό ανέρχεται σε 13%. Η Όλαφ μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης Ρέπλικα στην ουσία κατάσχεσε 113 ε, εκατομμύρια τσιγάρα που κατευθύνονταν στη χώρα μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ Όλαφ και ακτοφυλακών, καθώς και τις υπηρεσίε θελωνίων και εσόδων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο μας έτσι ώστε να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο ε, τσιγάρων. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τα stress test της 11, ε, οι 25 τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν. Ε, νέα από αυτές είναι Ιταλικές. Ε, έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Μέσα στα πλαίσια της ανάκαμψης της οικονομίας είδαμε ότι οι περισσότερες ταλικές τράπεζες χρειάζονται ενίσχυση δέκαδης ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή την ανακεφαλαιοποίηση θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, θα ήθελα να ρωτήσω πώς το τραπεζικό σύστημα θα ε, προωθήσει αυτή τη ροή και γιατί οι παράμετροι των τεστ αντοχής ήταν διαφορετικές σε σχέση με άλλες χώρες. Ίσως η Ιταλία δεν έχει το ίδιο ειδικό βάρος σε σχέση με άλλες χώρες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Σπέρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στο τέλος ε, της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου συζητούνται θέματα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και προβλήματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να πω ότι και τη Σλοβενία, την πατρίδα μου, εμείς ε, βλέπουμε τέτοια παραδείγματα παραβιάσεων δύο χρόνια καταδικάστηκε κάποιος ε, ο οποίος ε, ζήτησε ε, χρηματικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του. Η ποινή δεν θα εφαρμοστεί. Όμως υπάρχει ένας πολιτικός κρατούμενος στην Ευρώπη, ο οποίος ήδη εξέτησε 158 ημέρες από την ποινή που του επευλήθη. Ε, γι' αυτό χρειάζεται ε, να διαλευκανθούν αυτές οι υποθέσεις και ζητούμε τη βοήθεια της ε, Ευρώπης. Ο κύριος Σάιμον, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τελευταία φορά που ήρθα εδώ μίλησα για την εγγύηση για την νεολαία και την ε, αδυναμία της, ε, και την αποτυχία της Βρετανικής κυβέρνησης στο δεύτερο χρόνο που έτρεχε το πρόγραμμα να αντλήσει κεφάλαια. Τώρα θέλω να μιλήσω για τα χρήματα από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία ε, δεν δίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ανησυχούν, διότι οι τοπικές επιχειρηματικές συμπράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ε, έχουν την απαραίτητη διαφάνεια για να πάρουν τα κοινοτικά κονδύλια. Βέβαια, ε, η, ε, τα, τα κρίσιμα αυτά κεφάλαια δεν χρησιμοποιούνται και απευθύνω έκκληση και στην Κομισιόν και στο, στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Σιτς. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σκάνδαλο του Δικαστηρίου της Χάγης ε, για του εγκλήματα πολέμου. Είδαμε κι άλλο πλήγμα στην αξιοπιστία και το κύρος της Κροατίας. Ο κύριος Βέλσκο Μάριτς ε, υπηρετεί την ποινή του στη Σερβία, παρόλο που δεν ξέρουμε γιατί η σερβική δικαστική εξουσία είναι ε, αρμόδια και έχει δικαιοδοσία γι' αυτό. Διότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε κροατικό έδαφος ε, και θα έπρεπε να εκτίσει την ποινή του εκεί. Ε, ακόμα και όσοι εργάζονται σε ανθρωπιστικές αποστολές δεν μπορούν να τον επισκεφθούν ε, παρόλο που η υγεία του έχει υποσκαφθεί και δεν την χάνει της απαραίτητης ε, ιατρικής περίθαλψης. Ούτε μπορούμε και, και ε, υπήρχαν ήδη πάρα πολλά προβλήματα και στα στρατόπεδα ε, εγκλήστων και κατηγορουμένων για εγκλήματα πολέμου. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των ε, κατοίκων του Κερβίνιο. Ζουν ε, στο, στη βασική χώρα, αλλά ε, εντάσσονται στην Λεόν. Την προηγούμενη εβδομάδα τα μεγάλα ισπανικά κόμματα αρνήθηκαν τα δικαιώματα αυτών των κατοίκων. Και έτσι δυσχεραίνεται η καθημερινή τους ζωή. Πιστεύω ότι οι σοσιαλιστές και το Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να βρει ένα, ε, μία αντιμετώπιση, ενώ χρησιμοποιεί ένα νόμο του 14ου αιώνα. Εάν το πρόβλημα λοιπόν ε, ε, κινηθεί έτσι, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την αντιμετώπιση σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Το Νοέμβριο έγινε ένα δημοψήφισμα στην Καταλωνία όπου συμμετείχαν 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Δυστυχώς η κεντρική εξουσία δεν δέχτηκε την διενέργεια αυτού του δημοψηφίσματος και υπήρξαν πολλές απειλές. Το ίδιο ισχύει και στην ε, βασική χώρα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η αντιδημοκρατική στάση θα πρέπει να αναστραφεί και θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα ε, αυτοδιάθεσης των λαών. Αυτό είναι μια δημοκρατική αρχή και δεν μπορεί μια συγκεντρωτική αρχή να αρνηθεί αυτό το δικαίωμα. Sí, monsieur. La parole désormais, monsieur Terry Cabras. Terry Cabras. Oui. Pardon, Pardon. pour la prononciation. Perdón. Gracias, señora presidenta en Στις 9 Νοεμβρίου 2,5 εκατομμύρια πολίτες αποφάνθηκαν στα πλαίσια ενός εικονικού δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Η κυβέρνηση της Μαδρίτης αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα στο λαό. Αυτό είναι απαράδεκτο μία ευρωπαϊκή χώρα να μην επιτρέψει στους πολίτες να αποφανθούν ελεύθερα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθούν δημόσια για τα δικαιώματα, τα δημοκρατικά δικαιώματα των Καταλανών. Ο κύριος Ταμπουράνο. Ευχαριστώ. Στην Ελλάδα το ε, σύστημα, η δημόσια δέκο ηλεκτρισμού ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την ε, επίθεση της ΕΝΕΛ και επίσης υπήρξε μία προσπάθεια εξαγοράς Βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση όπου αυτή η Terna Corporation ε, είναι ε, μια αρχή ανταγωνισμού στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να πουλήσουμε, να πουληθούν τα ευρωπαϊκά asset για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση λιτότητας θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πώς η Ευρώπη θα επιλύσει ένα τέτοιο παράδοξο και πολλά άλλα που δεν μπορώ, επί των οποίων δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν έχω χρόνο. Ο κύριος Παπαδάκης. Η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα στην Ελλάδα με κριτήριο τα συμφέροντα του κεφαλαίου ετοιμάζουν προκλητικά νέα μείωση συντάξεων και την αύξηση του χρόνου κατοχήρωσης σύνταξης κατά πέντε έτη. Επίσης προωθούν την κατάργηση κοινωνικών πόρων που χρηματοδοτούν ασφαλιστικά ταμεία και επιδιώκουν να ενισχυθεί η λογική της ανταποδοτικότητας στο πνεύμα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. για να περάσουν αυτά και άλλα βάρβαρα μέτρα κλιμακώνεται ο αυταρχισμός οι διώξεις συνδικαλιστών ενώ συνεχίζουν να διατηρούνται επιστρατεύσεις απεργών. στο στόχαστρό τους έχουν το δικαίωμα στην απεργία για να αποδυναμώσουν την εργατική πάλη ενάντια στο κεφάλαιο. η έξαρση της καταστολής συνοδεύει την αντιλαϊκή πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης και κυβερνήσεων αποδεικνύει ότι αυτό που τρέμουν είναι τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό. απάντηση αποτελεσματική θα πάρουν στις 27 του νοέμβρη στη μεγάλη πανελλαδική απεργία για την κλιμάκωση της πάλης των εργαζομένων. κατά την 25η επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου βλέπουμε ότι πολλές υποσχέσεις για τις ανατολικές χώρες δεν έχουν πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία δεν έχουν ακόμη ξεριζωθεί πλήρως οι ολοκληρωτικές τάσεις γιορτάζουμε την ευρεία κοινωνική συνένεση που επιτεύχθηκε πριν από 25 χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμη φραγμοί στην ε, δημοκρατική λειτουργία και η Κομισιόν ήδη τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση του δικαστικού τομέα στη Σλοβενία γιατί καθοδηγείται από ανθρώπους που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα υπάρχει ακόμα το τείχος του Βερολίνου στη Σλοβενία. Μαρούσι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 Με την απελευθέρωση του κυρίου Σέσελ από το δικαστήριο της Χάγης ε, αυτό ακολουθήθηκε από τη δήλωση ότι η Σερβία πρέπει να έχει διέξοδο στη θάλασσα. Η Σερβία επίσης θέλει να είναι υποψήφια για ένταξη στην Ένωση αλλά δεν μπορεί η Ένωση να παραμένει σιωπηρή αν δεν διορθωθούν τα πράγματα στις ανατολικές χώρες. Ο κυρία Ζόργια Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Στη δύσκολη αυτή περίοδο όπου υπάρχουν εντάσεις μεταξύ θρησκειών και κοινοτήτων χρειάζεται το κοσμικό κράτος περισσότερο παρά ποτέ. Και νομίζω ότι είναι θλιβερό που θα έρθει αύριο ο Πάπας εδώ το, η Ολομέλεια δεν είναι το καταλληλότερο βήμα για τέτοιου είδους λόγους όταν παρουσιάζονται εδώ εκπρόσωποι θρησκευών και θρησκευτικών οργανώσεων. Εμείς είμαστε υπέρ της ανεξιθρησκείας αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός ορισμός του τι είναι κοσμικό κράτος που θα ήταν ο μόνος λογικός και δίκαιος τρόπος για να ζήσουν μαζί διάφορες κοινότητες. Εμείς δεν είμαστε εχθροί καμίας θρησκείας, αλλά υπέρ της ελευθερίας της συνείδησης. Ευχαριστώ. Κυρία Σελάνοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για την ενιαία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επιστολή στις 8 Αυγούστου προς ε, κάποιες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και αφορούσαν την κακή πρακτική γιατί πολλοί ε, πελάτες δεν μπορούν να βρουν την χαμηλότερη τιμή ανάλογα με το που διαμένουν. Στις 20 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε σχετικά με το τι κατάφερε να κάνει ε, οι εταιρείε ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούν να χρεώνουν διαφορετικά ανάλογα με τον τόπο διαμονής του πελάτη. Πρέπει όμως να το δικαιολογούν. Όμως αυτό οδηγεί σε διακρίσεις. παρόλα αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται εδώ δεν δικαιολογούνται. Και νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια παραβίαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, αρμόδια επίτροπο να καταπιαστεί με το θέμα αυτό. Χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όμως η Γερμανία αρνείται να καταβάλει στην Ελλάδα τις πολεμικές επανορθώσεις που επιδικάστηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη των Παρισίων το 1946 και ανέρχονται σε 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Επίσης αρνείται να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα παρότι και οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα η γερμανία αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα μου το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που επέβαλε το 1942 να της χορηγήσει η κατεχόμενη ελλάδα και το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 54 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. λόγω αυτού του δανείου διαλύθηκε η ελληνική οικονομία και πέθαναν από την πείνα πάνω από 600.000 Έλληνες. Επίσης 56.000 Έλληνες πατριώτες εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και 105.000 δολοφονήθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. όλα αυτά περιλαμβάνονται εδώ στη μαύρη βίβλο που εξέδωσε ο συνάδελφος μανώλης γλέζος. 162 δισεκατομμύρια ευρώ πλέον τόκων πρέπει να καταβάλει η Γερμανία για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αγγλικά. Ε, ένας ε, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλές διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών. Ε, καλές επικοινωνίες, οδικές, σιδηροδρομικές, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ε, Σλοβενία και την Κροατία να ολοκληρώσουν το την οδό Κόπαρ και από το Μάριμπορ στα κροατικά σύνορα επίσης και άλλη μια βασική αρτηρία γιατί αυτές οι τρεις είναι πολύ σημαντικές για την, τον τουρισμό, το εξαγωγικό εμπόριο και την επικοινωνία μεταξύ Ζάγκρεπ και Μάριμπορ. Και σε αυτά τα πλαίσια θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των έργων. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γλέζος, ένα λεπτό παρακαλώ. Η δημοκρατία στην Ελλάδα παραβιάζεται ασυστόλως όταν οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές όταν μάλιστα εξαιτίας της κρίσης υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα κυρίως νέων ανθρώπων το ελληνικό κράτος εμποδίζει όλους αυτούς να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα καθώς το κόστος μετακίνησης είναι απογορευτικό. τελικά θα ψηφίζουν μόνον οι πλούσιοι. γιατί η ελληνική κυβέρνηση κοφεύει στις εκκλήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και δεν δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους έλληνες να ψηφίζουν από τις χώρες διαμονής ενώ ψηφίζουν στις ευρωεκλογές; γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν σέβεται τα σχετικά ψηφίσματα του ευρωκοινοβουλίου και δεν εφαρμόζει παλιότερο σχετικό νόμο γιατί η ευρωπαϊκή ένωση δεν πιέζει την ελληνική κυβέρνηση ενώ κόπτεται για τη διάσωση των τραπεζών τελικά ποιος φοβάται ποιον σε αυτή την κρίση. Merci. Monsieur Ευχαριστώ. Στις 22 στα Κανάρια συνέβη κάτι το πολύ σοβαρό. Η Greenpeace στην ουσία διαδήλωνε κατά της Ρεψόλ αλλά δυστυχώς της ε, επιτέθηκε η ακτοφυλακή. Αυτό αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρήση του στρατού δημιούργησε μεγάλη ανασφάλεια στο, στους πολίτες. Επίσης έγιναν και σοβαρές ζημιές. Γι' αυτό θα θέλαμε να ε, απελευθερωθούν οι κρατούμενοι και να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να δηλώνουν όταν το επιθυμούν. Η κυρία Εύη. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών ισχύει από το γύρο της Ντόχα. Θεωρήσαμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε καλύτερες τεχνολογίες. Όταν το διοξίδιο του άνθρακα στήχιζε πολύ περισσότερο, στο το 2009 ψηφίστηκε αυτό το σύστημα, αλλά μιλάμε για κόστος που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ε, επιτρέψουμε τον παρασιτισμό των χρηματιστών. Ήρθε η ώρα να προωθήσουμε συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά το σύστημα ETS. Η κυρία Βόζεμπεργκ τα τελευταία χρόνια στην ευρώπη μεγάλο μέρο των συμπολιτών μα διαβιεί κάτω από το όριο τη φτώχεια, εξαιτία των πολιτικών λιτότητα και μέτρων δημοσιονομική προσαρμογή που εφαρμόζονται σε πολλά κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 120 εκατομμύρια ευρωπαίοι ζουν κάτω από αυτό το καθεστώ, σύμφωνα με στοιχεία τη eurostat το. 2013. η χώρα μου η ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση των χωρών τη Ευρώπη, με υψηλότερο ποσοστό φτώχεια ενώ η ανεργία ξεπερνά το 27% το γεγονός αποκαλύπτει το βάθος της κρίσης με τέσσερα εκατομμύρια περίπου έλληνες άπορους και κοινωνικά αποκλεισμένου, να αδυνατούν να καλύψουν τα προστοζήνα αναγκαία διότι μεταξύ άλλων 230.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν, θέσεις εργασίας χάθηκαν και αυξήθηκαν δραματικά τα φαινόμενα εξαθλίωσης κοινωνικής. Η Ευρώπη πρέπει εδώ και τώρα να αντιμετωπίσει την εξάπλωση της φτώχειας αποτελεσματικά, να ακολουθήσει στρατηγική μακρόπνοου χαρακτήρα με στόχο και σκοπό τη σταδιακή αποκατάσταση του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων, ιδίως στις χώρες που το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο κυρία Γκραπίνη για ένα λεπτό. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ελευθεροτυπίας στην ναι. χώρα μου. Ο κύριος ε, Βοικουλέσκι, Βοικουλέσκου ήρθε σε επαφή με τον αδελφό του πρώην Προέδρου Προέδρου του κυρίου Μπασέσκου και χειραγώγησαν τον τύπο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την πραγματογνωμοσύνη όπως προωθήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο Νταν Βοικουλέσκου είναι επικεφαλής ενός πολύ μεγάλου τράστα. Επίσης ε, ενεπλάκησαν και άλλα ε, μέρη τα οποία δεν είχαν σχέση με την υπόθεση. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τύπος βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και δεν ξέρω πώς θα επιβιώσει. Σάνι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, οικονομική κυρίως. Ε, πρόσφατα εγκρίναμε συμφωνία σύνδεσης ε, με την Ουκρανία, που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε κάποιες ευθύνες. Δεν είναι όπως η συμφωνία σύνδεσης ε, μεταξύ Ουγγαρίας τώρα ε, υπάρχει πρόβλημα ενεργειακού εφοδιασμού και από την Ευρώπη δεν τονίστηκε αρκετά το θέμα, δηλαδή να ε, παρασχεθεί η απαραίτητη υποδομή στην Ουκρανία και στις άλλες συνδεδεμένες χώρες. Ε, νομίζω ότι είναι καλύτερα να δράσουμε από τώρα προληπτικά παρά αργότερα για να, όταν θα έχει ξεσπάσει το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βαλίνα. ευχαριστώ αύριο θα ε, πανηγυρίσουμε και θα γιορτάσουμε την ημέρα ισότητας των δύο φύλων. Το 52% του πληθυσμού είναι γυναίκες και ο οργανισμός ε, ίσων δικαιωμάτων δείχνει ότι 62 εκατομμύρια γυναίκες υφίστανται ε, βία, πράξεις βίας από τους άνδρες. Ο ίδιος ο οργανισμός μιλά για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν μπορεί να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα θέλαμε όλα τα κράτη να ψηφίσουν την συνθήκη της Ισταμπούλ. Και να λάβουμε υπόψη τα θύματα παντού και στην Ισπανία που είναι πολλά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απαλείψουμε αυτή τη μάστιγα. Ο κύριος Φερνάντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη θα ασχοληθεί με το επενδυτικό, επενδυτικό πρόγραμμα της Επιτροπής Juncker. Έγινε λόγος για την χρηματοδότηση 300 δις. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα επιλεγούν τα προγράμματα και πώς θα γίνει η κατανομή των διαφόρων ε, προγραμμάτων. Στην Ισπανία μάθαμε ότι θα υπάρξουν επενδυτικά σχέδια χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αυτόνομες περιοχές. Θα ήθελα ο κύριος Τίμερμαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη πολύ προσεκτικά μία διαδικασία ε, διαφανούς επιλογής των προγραμμάτων. Ο κύριος Τόκες. Ρωμανιά, 25 χρόνια πριν από με a Ceausescu δικτατούρα az idei jubileum legszebb ajándéka klaus johannis demokrata liberális στην ε, ε, Ουγγαρία ε, τα προηγούμενα 25 χρόνια ε, ήλθαν ε, πολλοί κομμουνιστές σε ανώτερα αξιώματα. Ε, αυτό θα έπρεπε να αλλάξει. Στις εκλογές είδαμε το λεγόμενο αποτέλεσμα αντίκτυπο Ομπάμα. Είχαμε την τιμή άρα παλιά, τώρα η Τρανσιλβανία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή. Οι Ούγγροι και οι Γερμανοί ε, διώχθηκαν από τον Τσαουσέσκο μαζί με τους ε, Ρουμάνους συμπατριώτες τους. Όλοι τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής. Την ε, περασμένη Παρασκευή όλη η Λετωνία τίμησε τη μνήμη της τραγωδίας της ζολιτούντες στη Ρήγα ε, στις 21 Νοεμβρίου του 2013 το ένα σούπερ μάρκετ κατέρευσε και 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ε, ήταν ε, το μεγαλύτερο ατύχημα στην ιστορία της Λετωνίας και η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ανατολική Ευρώπη τα προηγούμενα 30 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πέθαναν λόγω τρομοκρατικού πλήγματος ή φυσικής καταστροφής, ε, αλλά μέσα σε ένα κατάστημα σε εποχή ειρήνης. ακόμα κανείς δεν έχει διωχθεί ένα χρόνο μετά. Η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης δεν ξέρουν ποιος έφτεξε. Ακόμα η αστυνομία και ο εισαγγελέας δεν έχουν τελειώσει τις, ε, τις έρευνες ε, και σταμάτησαν να καταβάλλονται κοινωνικά επιδόματα στα, ε, στις οικογένειες των θυμάτων. κύριος Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω για την αλλαγή της ώρας. Εδώ και μερικές δεκαετίες άρχισε να, να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο στην Ευρώπη με βασικό στόχο τη δια... εξοικονόμηση ενεργείας. Αλλά τώρα με τις καινούργιες εξελίξεις στην οικονομία και στη γεωργία και στις μεταφορές δεν είναι πλέον απαραίτητο να γίνεται. Και διαπιστώθηκε ότι ό,τι εξοικονομούμε το πρωί το χάνουμε το βράδυ και πολλές χώρες και στη Λατινική Αμερική και αλλού το παράτησαν το σύστημα. Οι πολίτες μας ε, δεν το εγκρίνουν επίσης γιατί διαταράσει τον ύπνο τους και γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να συζητήσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεπαρτέλ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, Τα στοιχεία για την ανεργία των νέων μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει σίγουρο μέλλον για τους ε, νέους μας. Ως νέα ευρωβουλευτής ε, κατανοώ το πρόβλημα των ε, νέων. Η κοινωνία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Οι νέοι μας χρειάζονται, εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε Έχουμε 5,3 εκατομμύρια ε, νέους χωρίς εργασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το μέσο εγγύησης των νέων και να προβούμε σε επενδύσεις για, τον ε, μέλο για το μέλλον των νέων μας. Θα πρέπει να προωθήσουμε διεθνικά σχέδια και προγράμματα για τους νέους. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ε, νέους ε, να μπορέσουν να ανταποκριθούν, να αποκτήσουν πείρα και να είναι δραστήριοι στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Έτσι κλείνει η συνεδρίασή μας. Τη 3η 25 ε, Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση και στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.